Vamos a Ξεκινήσουμε την ψηφοφορία. Το πρώτο σημείο είναι η έκθεση Καζίνη για τη διαθεσμική συμφωνία Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τη Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Μία μόνο ψήφος. Ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχέ εγκρίνεται. Να περάσουμε την αριθμητική σύνθεση των δικαιολογικών αντιπροσωπείων και άλλων αντιπροσωπείων. Έχουμε την πρόταση συνολικά υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Τώρα, έκθεση Τσέσκοβα. Απαλλαγή 2011 του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του Συμβουλίου των Υπουργών. Δεν υπάρχουν τροπολογίες. Ψηφίζουμε. Υπέρ. Κατά Αποχές. Εγκρίνεται. Να ψηφίσουμε τώρα το ψήφισμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συνάδελφοι, όπως ξέρετε, Έχουμε τώρα ένα δικαιωμένο επισκέπτη που είναι ο πρόεδρος της Ενεγάλης. Βεβαίως, ο πρόεδρος της Ενεγάλης. Θα διακόψουμε την ψηφοφορία για να κάνουμε την επίσημη συνεδρίαση. Αντί να ψηφίσουμε λοιπόν την έκθεση Τζανόνι, η οποία θα μας πάρει πολύ χρόνο, άρα θα έχουμε δυσχέρειε με το χρονοδιάγραμμα, θα ψηφίσουμε άλλες εκθέσει που είναι πιο σύντομες και η έκθεση Τζανόνι θα ψηφιστεί μετά την επίσημη συνεδρίαση. Θα περάσουμε στην έκθεση Harbour. για τα σκάφη αναψυχής και ατομικά σκάφη. Έκθεση Harbour. Ψηφίζουμε το μπλοκ 1 τροπολογιών. Ονομαστική άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται το μπλοκ 1. Να ψηφίσουμε τώρα την πρόταση της Επιτροπής. Ονομαστική άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Να ψηφίσουμε το νομοθετικό ψήφισμα. Ονομαστική άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Τώρα να περάσουμε στην έκθεση Βερνιού για την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων. Πρώτα το μπλοκ αριθμός 1, ονομαστική άρχεται. Α, το πρώτο τμήμα, το πρώτο τμήμα. Είναι ε, απλή ψηφοφορία. Το πρώτο τμήμα του πρώτου μπλοκ. Ποιοι είναι υπέρ παρακαλώ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τώρα ψηφίζουμε το δεύτερο τμήμα. Ονομαστική άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. να ψηφίσουμε τώρα την πρόταση της Επιτροπής Ονομαστική Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Και τώρα, πριν ψηφίσουμε το νομοθετικό ψήφισμα, να ψηφίσουμε την τροπολογία 161 υπέρ παρακαλώ κατά αποχές εγκρίνεται και τώρα να ψηφίσουμε το νομοθετικό ψήφισμα ονομαστική άρχεται πέρας εγκρίνεται τώρα θα ψηφίσουμε την έκθεση Bauer για τη Συμφωνία Ένωσης Αρμενίας για τις προξενικές θεωρήσεις υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Περνάμε τώρα στην άλλη έκθεση Bauer Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Αρμενίας για ε, παράνομους ε, κατοίκους. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τώρα για επιτρεπόμενη χειρισμοί υγείας για τρόφιμα δεν έχουμε τροπολογίες ε, πρέπει να έχουμε ειδική ε, πλειοψηφία. Παρακαλώ, ποιοι είναι υπέρ, σηκώστε ε, το χέρι σας παρακαλώ. Κατά. Λοιπόν, πρέπει να ελέγξουμε. Ηλεκτρονικά έρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. Τώρα να περάσουμε τρόφιμα και προϊόντα ζωικής προέλευσης Ψηφίζουμε την πρόταση ψηφίσματος και πάλι χρειαζόμαστε ειδική πλειοψηφία υπέρ. Κατά. Αποχές. Πρέπει να κάνουμε έλεγχο. Άρχεται. Άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. Τώρα να περάσουμε για τις διαπραγματεύσεις με την Κίνα. Λοιπόν, οι ένα και έξι είναι ταυτόσιμες, από κοινού ονομαστική άρχεται. Πέρας. Απορρίπτονται. Παράγραφος 17, δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα, ονομαστική άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 2. Ονομαστική άρχεται. Πέρας εγκρίνεται. Οπότε περνάμε στην παράγραφο 26 τρία τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Και τρίτο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 36, τροπολογία 3, ονομαστική άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 7, ονομαστική άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. Παράγραφος 41. Πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Ονομαστική. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Να ψηφίσουμε την τροπολογία 4. Ονομαστική. Άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. Παράγραφος 42, δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα, ονομαστική άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 5. Ονομαστική άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. Οκτώ ονομαστική άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. Και τώρα ψηφίζουμε την παράγραφο 43, τρία τμήματα. Το πρώτο τμήμα υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά αποχές Λοιπόν, ωραία, ηλεκτρονικός έλεγχος για το δεύτερο τμήμα της παραγράφου 43. Πέρασε. Εγκρίνεται. Το τρίτο τμήμα δεν το ψηφίζουμε, έχει αποσυρθεί. Τώρα να ψηφίσουμε συνολικά την πρόταση. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Περνάμε στο επόμενο θέμα. Ωραία. Έχουμε χρόνο για άλλη μια ψηφοφορία ε, σχέση με την Ταϊουάν. Η παράγραφος 1-2 τμήματα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 1 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται να ψηφίσουμε την παράγραφο 4 τώρα υπέρ κατά λοιπόν να ελέγξουμε ηλεκτρονικά άρχεται παράγραφος 4 πέρασε εγκρίνεται να ψηφίσουμε τώρα την τροπολογία 2 ονομαστική άρχεται Πέρας. Απορρίπτεται. Να ψηφίσουμε λοιπόν τώρα την παράγραφο 4, λέει ο Πρόεδρος, ε, ε, ε, ονομαστική άρχεται. Με συγχωρείτε, παράγραφο 14. Ψηφίζουμε την παράγραφο 14 ονομαστική. Πέρας. Εγκρίνεται. Ψηφίζουμε συνολικά την πρόταση. Άρχεται. Συγγνώμη, υπέρ, κατά, αποχές. Εγκρίνεται. Ωραία. Και τώρα θα διακόψουμε τις ε, ψηφοφορίες για την επίσημη συνεδρίαση. Άλλη μία. Εντάξει, ωραία. Να ψηφίσουμε λοιπόν Άλλη μία. Θέλετε άλλη μία. Λοιπόν, άλλη μία. Η κυρία Λίχτενμπεργα. Παρακαλώ. Α, αγαπητοί συνάδελφοι, πριν αρχίσετε να με σφυρίζετε, ακούστε τι έχω να πω. Χθες τη συζήτηση για τους χρόνους πτήσης και ανάπαυσης για τους πιλότους και το πλήρωμα καμπίνας μας είπε ο Επίτροπος Κάλλας ότι υπάρχουν νέες προτάσεις και μας τις υπέβαλε που είναι αποτέλεσμα διαπραγματεύσεων μεταξύ αυτού και το Συνδικάτο των Εργαζομένων στον τομέα αυτό. Αυτές οι προτάσεις αλλάζουν τη βάση συζήτησης που είχαμε στην Επιτροπή αλλά αυτό το είπε με γενικό τρόπο. Δεν ξέρουμε τι ακριβώς περιέχουν αυτές οι αλλαγές και ποιο είναι τώρα το περιεχόμενο της πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το ψήφισμα που πρόκειται να ψηφίσουμε τώρα απορρίπτει την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Διότι εμείς εργαστήκαμε με βάση την προηγούμενη πρόταση. Γι' αυτό πιστεύω ότι ένα κοινοβούλιο πρέπει να γνωρίζει τι ψηφίζει. Γι' αυτό σας παρακαλώ να αναβάλουμε την ψηφοφορία ούτω ώστε να έχει το Κοινοβούλιο την ευκαιρία να μελετήσει τις προτάσεις του Επιτρόπου να τις λάβει γραπτός και να τις συζητήσει. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Λίχτεμπεργκ, βάσει του κανονισμού η πρότασή σας μπορεί να έχει έναν αγωγητή υπέρ και έναν κατά. Υπάρχει κάποιος που θέλει να υποστηρίξει την πρόταση της κυρίας Λίχτεμπεργκ. Όχι. Κάποιος θέλει να μιλήσει κατά. Ναι, όχι. Κύριε Πρόεδρε, είμαι υπέρ με πολύ σκεπτικισμό αντιμετωπίζω τον κανονισμό που μα είπε η Κομισιόν. Δεν ξέρω αν είναι καλό. Αν έχουμε μια δυνατότητα να τον βελτιώσουμε, ούτω ώστε να υπερψηφίσουμε, να αξιοποιήσουμε αυτή την πρόταση και να έχουμε το χρόνο να την αξιοποιήσουμε. Ευχαριστώ. Κάποιο αγωγητή κατά. Όχι. Ο κύριος Σπερώνη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πιστεύω ότι στη φάση που βρισκόμαστε μια ψηφοφορία από πλευράς Κοινοβουλίου για την πρόταση ψηφίσματο θα διευκολύνει, μόνο θα διευκολύνει τι θέσει μα έναντι του Συμβουλίου και τη Επιτροπή. Ωραία, λέει ο Πρόεδρο. Ψηφίζουμε τώρα την πρόταση Λίχτεμπεργκ. Ποιοι είναι υπέρ, όσοι είναι υπέρ θα ψηφίσουν υπέρ, όσοι είναι κατά θα ψηφίσουν κατά. Ψήφι υπέρ της πρότασης της κυρίας Λίχτεμπεργκ. Ψήφι κατά θα γίνει ηλεκτρονικός έλεγχος. Η ηλεκτρονική ψηφοφορία άρχεται η ψηφοφορία. Σε cierra la votación. Πέρας ψηφοφορίας. Η πρόταση της κυρίας Λίχθενμπεργκ απορρίφθηκε. Ψηφίζουμε τώρα τις απαιτήσει για τις αεροπορικές δραστηριότητες με ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Σε Πέρας ψηφοφορίας. Η πρόταση απορρίφθηκε. Ωραία. Τώρα θα διακόψουμε την συνεδρίαση ούτω ώστε να ακούσουμε τον πρόεδρο της Ενεγάλης και κατόπιν θα συνεχίσουμε με, τα εκκρεμή, με τις